Good morning, friends. Uh, we'll start with the voting session <clears throat> immediately. I hope you have put your... ξεκινάμε αμέσως με την ε, ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε φέρει τις ε, κάρτες ε, ψηφοφορίας. Για να είστε έτοιμοι να πατήσετε το κουμπάκι. Ωραία. Περιμένουμε τον κύριο Λέναρ και τον κύριο Μπέκερ. Και ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία. Και είναι και ένα ερώτημα προς την Κομισιόν, προς τον κύριο Χέντελ, ονομαστική ψηφοφορία για το ΕΤΠΟΥ και την Νόκια στην Φιλανδία. Είναι ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ και τους σοσιαλδημοκράτες. Ένας παραπάνω από τους σοσιαλδημοκράτες. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. 43 υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Λαμπάγιοβα. Mm. Uh, Madame Λαμπάγιοβα. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, ξέχασα την κάρτα μου, αλλά είμαι εδώ εν πάση περιπτώσει. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι, πολλοί δεν έφεραν τις κάρτες τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Περνάμε στο επόμενο θέμα. ερώτηση για προφορική απάντηση Χέντελ για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσώπων για την Διαβίου Μάθηση. Και ξεκινάμε με την συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Άρα, η τροπολογία 1, 2, 3 καταπίπτουν, 4 καταπίπτει, Α, όχι, την 4 θα ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία καταπίπτει, καταπίπτει. Πάμε στη 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το παρηθεύσουμε νομίζω. 15. Άρχεται η ψηφοφορία. και πέρας και απορρίπτεται με 26 ψήφους 16 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε και αυτή να έρχεται η ψηφοφορία πέρας και καταπίπτει είναι δύσκολα τα πράγματα. Άλλοι δεν έχουν την κάρτα, φέρει. Η κυρία Παλώμα ήταν υπέρ, η κυρία Λαμπάγιοβα ήταν κατά. Οπότε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Άρα απορρίπτεται. Περνάμε. στην 17 υπέρ. Κατά αποχές να το επαληθεύσουμε. Και πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική ερώτηση όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. με 47 ψήφους υπέρ εγκρίνεται και τρεις αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή. Ε, δεν είναι εδώ, αλλά θα το μεταφέρετε φαντάζομαι. Και περνάμε Ε, σχέδιο ψηφίσματος, συμβαστική β υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Συμβαστική γάμα, τροπολογία 52, 52 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Συγγνώμη. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική γάμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και δεκτή. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε την 75 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας και απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 77 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 78 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79, την επαληθεύουμε, άρχη η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται με 10 ψήφους. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές. Εγώ νομίζω ότι έγινε δεκτή. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Δεκτή με 29 ψήφους. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται επαληθεύουμε την 84. Συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 94 υπέρ κατά αποχές. Εγώ νομίζω δεκτή. 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 96 υπέρ κατά αποχές δεκτή 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές δεκτή 99 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 99 να έρχεται η ψηφοφορία πέρας Δεκτή. 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ Κατά. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 111. Για να είναι απόλυτα σαφές. Ωραία. Πέρας. Σας ευχαριστώ. Επικρατεί σύγχυση. Εγώ δηλαδή μπερδεύτηκα. Ήσασταν τόσο ενωμένοι που νόμιζα ήταν λάθος. Συμβαστική G υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 119 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 120 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές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 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Με 37 ψήφους. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά νομίζω θα πρέπει να ελέγξουμε γιατί 12 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και απορρίπτεται κατά μία ψήφο 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε για τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται κατά μία ψήφο. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 17, καταπίπτει, 18 υπέρ, α, καταπίπτει επίσης, όχι, όχι, ψηφίζουμε τη 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική A υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 22 όχι, όχι. Ψηφίζουμε την 27. 27. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήταν η 27 και 28. Γιατί ήταν ταυτόσημες, άρα ε, ξαναψηφίζουμε τις 27 και 28. Υπέρ 27-28. Κατά αποχές απορρίπτονται. 29 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Εγκρίνεται με 31 ψήφους. 34. 34 καταπίπτει 31 υπέρ. Κατά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 και εγκρίνεται με 38 ψήφους. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίσουμε το σχέδιο όπως έχει τροποποιηθεί και άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. εγκρίνεται με 50 ψήφους υπέρ. Τρεις κατά. Και να συγχαρούμε τον κύριο Χέντλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος.

Ε, συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη πρόταση κανονισμού για τους απάτριδες ε, ή εκείνους που δικαιούνται επικουρική προστασία και λοιπά και λοιπά. Αρχίζουμε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 121 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Α, να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε την 128. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Σας ευχαριστώ. 127, 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά. Εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε για την 133 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε την 137 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Τώρα είμαστε εντάξει. Ε, απορρίπτεται κατά μία ψήφο. 138 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 141 και 142 καταπίπτουν 143. Ψηφίζουμε? Ναι, ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16, καταπίπτει, όχι, όχι, ψηφίζουμε τη 16 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 16, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 35 υπέρ. Εγκρίθηκε. 144 ψηφίζουμε υπέρ Η ειδική λένε ότι ψηφίζουμε. Ωραία, ας ψηφίσουμε. 144 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 147, άρχεται η ψηφοφορία και τώρα πέρας και απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 τι κάνουμε, την ψηφίζουμε, ωραία. Υπέρ, κατά αποχές και εγκρίνεται. 149. Καταπίπτει. Συμβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε λοιπόν τη συμβαστική τοπολογία H, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται λοιπόν. Οπότε θα ψηφίσουμε από τις 150. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Οπότε στις 18 και 151. Ψηφίζουμε δηλαδή από κοινό για αυτές τις δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ας ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά. 18 και 151. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται λοιπόν. Διαφορά τριών ψήφων. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ας την ελέγξουμε λοιπόν. 153. Αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε την 159. Λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με διαφορά τριών ψήφων. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ 173 διορθώνει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 και 179 υπέρ κατά αποχές ας τις ελέγξουμε 178 λοιπόν και 179 από κοινού άρχεται η ψηφοφορία πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 180 υπέρ κατά ή μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας σίγουρα απορρίπτεται. 181 Αποκινούμε την 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ, ή μάλλον καταπίπτει 186, συμβαστική τροπολογία L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 188 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 189 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 190 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 πίπτη οπότε πάμε στην 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και είναι ψήφος για την 199 200 και 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 203 καταπίπτει περνάμε στην τροπολογία 25 ή μάλλον από κοινού 25, 204, 205, 206, 207 υπέρ, κατά, αποχές εκρίνονται. Αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται λοιπόν με 36 ψήφους υπέρ, 208 υπέρ, κατά, ποιες απορρίπτεται. Η 209 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην 211. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως πρέπει να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν, την 26, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται λοιπόν με 28 ψήφους κατά 212 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 214. Α, όχι, να ελέγξουμε τη 213 ηλεκτρονικά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Πράγματι, απορρίφθηκε. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε τη 215 για να είμαστε σίγουροι. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε πράγματι. 216 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 223 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ, κατά αποχές ας ελέγξουμε την 225 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται λοιπόν με διαφορά δύο ψήφων 227 καταπίπτει οπότε πάμε στην 228 αποκινούμε τη 229 ψήφι Πέρα κατά αποχές απορρίπτονται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 231 υπέρ καταπίπτει 231 και η 232 καταπίπτει οπότε περνάμε στην τροπολογία 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία B υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 καταπίπτει 57 και η 58 καταπίπτει περνάμε στην 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 Αποκινούμε την 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρινώνται. Συμβαστική τροπολογία D, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 και τροπολογία 77 καταπίπτουν περνάμε στην τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 85 καταπίπτει πάμε στην 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 καταπίπτει όχι δεν καταπίπτει 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές για να την ελέγξουμε Πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας. Πράγματι σας ευχαριστώ. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την συμβαστική τροπολογία F. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Οπότε 96 υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε τα 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Όμως αναφέρεται εδώ ότι καταπίπτει αν έχει εγκριθεί η συμβαστική τροπολογία Ή και η συμβαστική τροπολογία Ή εγκρίθηκε πράγματι. Πρόεδρος, έχει γίνει ένα λάθος ο κατάλογος ψηφοφορίας στο voting list. Οπότε, ας επαναλάβουμε την ηλεκτρονική μας ψηφοφορία για την τροπολογία 96. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Άρα λοιπόν εγκρίνεται. Περνάμε στην 14 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει 14. Πηγαίνουμε λοιπόν στην 101, τοπολογία 101, στον αδελφο Λορανά. Υπέρ λοιπόν, Είμαστε στη σελίδα 18 λοιπόν του voting list. Άρα λοιπόν, αφού υπερψηφίσαμε την 96, όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν έως την 101, την οποία θα ψηφίσουμε τώρα. Τροπολογία λοιπόν του συναδέλφου Ρολά ψήφι Κατά, αποχές, Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην Άρα λοιπόν εγκρίθηκε η 101. Περνάμε λοιπόν στην 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου έκθεσης, ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν, άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρας και εγκρίνεται με 41 ψήφους υπέρ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εισηγητή για όλη τη δουλειά που έχει κάνει εδώ. We uh, uh, Συνεχίζουμε με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. 11. 11 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική F υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ελέγχουμε, ελέγχουμε την 33, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και απορρίπτεται κατά δύο ψήφους 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτεται ελέγχουμε την 45 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται κατά μία ψήφο. D υπέρ, κατά της συμβαστικής αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 49 ε, καταπίπτει, άρα πάμε στη συμβαστική K υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ Α, με συγχωρείτε, 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 στις αιτιολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε στη γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί και άρχεται η ψηφοφορία και κλείνει και εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ και 3 κατά και ευχαριστούμε τον εισηγητή. Μετά έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Is it a difference? This 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Edouard Martin. Mm. Okay. Uh, when it comes to the... Uh, Μάλιστα. Λοιπόν, κανόνες που αφορούν τον προπολογισμό της Ένωσης, όπως ξέρετε, στο Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης έχει αναβληθεί η ψηφοφορία για τις 15 Μαΐου για το Στρασβούργο, οπότε τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες και περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι το πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης, δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, ε, χρεποποίησης και απαλλαγής. Λοιπόν, παρακαλώ οι συζητήσει ε, εκτός της αιθούσης. Και θα δώσω σύντομα τον λόγο στον εισηγητή Εντουάρτ Μαρτάν. Παρακαλώ, χαμηλόφωνα. Γιατί έχουμε ένα σημαντικό θέμα στη μερίσια διάταξη. Με συγχωρείτε, Ρωσιά. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μαρτάν. Έχετε τον λόγο. Mr. Martin. Μαρτάν. Oui, oui, merci, Madame la Présidente, mais j'attends Ευχαριστώ. Περιμένω να επικρατήσει ησυχία, γιατί φαίνεται ότι το θέμα δεν ενδιαφέρει πολλούς, άρα συνεχίσουν τις συζητήσεις εκτός αίθουσας. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για μία γνωμοδότηση. Η Γιούρη είναι υπεύθυνη επί της ουσίας. Η προθεσμία για τις τροπολογίες ήταν η 10η Μαΐου στις 12. Επειδή η Γιούρη χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο, προτείνω να παρατείνουμε στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, έτσι ώστε και άλλες ομάδες να έχουν χρόνο. Σε σχέση με την πρόταση αυτή της πρότασης νομοθετικού περιεχομένου αφορά τα προσόντα των εργαζομένων σε μια επιχείρηση οι οποίοι είναι πιστωτές ε, όπως και κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και αυτή είναι η θεώρηση της Επιτροπής. Άρα μιλάμε και για ένα ε, σκέλος αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης στην οποία θα πρέπει να δούμε κατά πόσο συμμετέχουν ή όχι οι εργαζόμενοι. Ορίζουμε λοιπόν τον ε, πιστοτή και τον θεωρούμε ταυτόσιμο με τον καταναλωτή. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε σε επίπεδο κατανάλωσης πώς ισχύουν όλα αυτά ορίζοντας τους εργαζόμενους ως καταναλωτές, τους θεωρούμε παράλληλα και πίστοτες. Αυτή είναι η κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να ορίσουμε την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης, που, όπου δεν υπάρχει μόνο συμβατική σχέση μεταξύ επιχειρήσεων ε, κεφαλαιοδοτικών οργανισμών και εργαζόμενων. Θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε για μια συλλογική εργασία και υπ' αυτή την έννοια ο εργαζόμενος δεν ταυτίζεται με αυτή την προηγούμενη κατηγορία. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι λοιπόν να τύχουν αναγνώρισης και να υπάρχει ένα σύστημα προειδοποίησης εάν η οικονομική κατάσταση είναι δυσχερής και εάν υπάρχει θέμα αναδιάρθρωσης επιχείρησης θα πρέπει να διαδραματίζουν τον ίδιο ε, ρόλο με τις πιστοτικές αρχές. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των μέσων για την ανάλυση της κατάστασης επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ενδυνάμει κατάσταση των συνταξιούχων τη στιγμή που υπάρχει ένα συνταξιοδοτικό σχήμα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις προδιαγραφές της οδηγίας. Η Επιτροπή χαίρεται για τις θετικές επιπτώσεις του δικαιώματος στην πληροφόρηση, αλλά το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να είναι πραγματικό. Ε, αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το άρθρο 27 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων μιλά για το δικαίωμα πληροφόρησης των εργαζομένων στην επιχείρηση. Γι' αυτό θα πρέπει, ε, εάν γίνει μία ε, προγενέστερη αναδιάρθρωση, να υπόκειται σε κοινωνικό διάλογο, γιατί δεν θα πρέπει να πλήτεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στην αναδιάρθρωση. Τέλος, οι τροπολογίες ε, ορίζουν τέσσερα από τα οκτώ σημεία της μελέτης αντικτύπου, δηλαδή την ε, δυνατότητα αναδιάρθρωσης, την, και επίσης την δυνατότητα πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης και φυσικά καλύτερη δυνατότητα ανα, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, αφαιρεγγιότητας και απαλλαγής στην περίπτωση, και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις διαβουλεύσεις. Είμαι στη διάθεση των σκιωδών για να βελτιώσουμε το κείμενο. Thank you. Uh, I'll now give the floor to Madam... Uh, Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Λόπες Φοντανέ. Έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης που μόλις μας παρουσίασε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε εκ των υστέρων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασίζεται με θέματα απασχόλησης, σε θέματα απασχόλησης. Τώρα, ε, ως προς το θέμα των πιστωτών και των οφηλετών θα πρέπει να δούμε πώς έχει η νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού υπάρχει αφαιρεγγιότητα και να δοθεί μία ε, δεύτερη ευκαιρία, ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες καλής πίστης. Αυτό ε, σημαίνει δηλαδή ότι η αναδιάρθρωση θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Άρα η πρόταση της Επιτροπής είναι μία εξισορροπημένη πρόταση που ορίζει ορισμένες πτυχές τελικής εναρμόνισης. Μιλάμε για προληπτική δηλαδή αναδιάρθρωση και τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε υγιείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για εκείνους που, δουν, που δρούν διασυνοριακά δηλαδή που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα ελεύθερης εγκατάστασης. Ε, υπ' αυτή την έννοια θα κινηθούν και οι τροπολογίες μου. Ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις θέσεις εργασίας και τη διατήρησή τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, λειτουργικότητα των επιχειρήσεων και να μην διαλύονται οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά σημεία που με βρίσκουν ε, σύμφωνοι με τον εισηγητή, αλλά επειδή μιλάμε για μια ειδική κατηγορία, δηλαδή τους εργαζόμενους, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε υπόψη το ζήτημα στην ολότητά του και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα διαβούλευσης των εργαζομένων με τους εργαζόμενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προβαίνουν σε μία προειδοποίηση των ευρωπαϊκών αρχών εάν η αναδιάρθρωση έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζομένους. Επίσης θα μπορούσαμε να προβούμε σε μια πραγματογνωμοσύνη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αλλά αυτό θα μπορούσε όμως να είναι δαπανηρό και θα παρατείνει τις προθεσμίες και ειδικά για τον οφιλέτη. Στην τροπολογία 2 μιλάμε για την ε, προληπτική αναδιάρθρωση, το οποίο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει συρρήκνωση μισθών θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία των επιχειρήσεων, γιατί στη δική μου περιφέρεια το 2013 η General Motors αντιμετώπισε προβλήματα, φτάσαν σε μια συμφωνία οι εργαζόμενοι με την επιχείρηση με τα συνδικάτα δηλαδή επήλθε συμφωνία και διατηρήθηκαν όλες οι θέσεις εργασίας. Πολλές φορές είναι πολύ καλό τα συνδικάτα να προβούν σε διαβουλεύσεις και για να φτάσουμε σε μια μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το συνταξιοδοτικό σχήμα. Εν μέρη μου απάντησε ο εισηγητής και θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σεντάνσκα έχει τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Να ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και χρεοκοπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο 200.000 επιχειρήσεις ε, κλείνουν κάτι το οποίο σημαίνει 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις κάτι το οποίο θα σήμαινε 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε πως είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ε, καταστάσεις ε, χρεοκοπίας στις επιχειρήσεις σχετίζεται με την κύκλικη πορεία της οικονομίας, κάποιους κραδασμούς ή έντονο ανταγωνισμό στην αγορά. Γνωρίζουμε ότι στα κράτη-μέλη έχουμε νομοθεσία που αντιμετωπίζει το ζήτημα κυρίως για διαδικασίες αναδιάρθρωσης η οποία φροντίζει και για προστασία των δανειστών. Πέρα από αυτό υπάρχει και μια σπίδα προστασίας για τους εργαζόμενους με βάση το άρθρο 27 της ε, Χάρτας των Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην διαβούλευση και στην παροχή πληροφόρησης και κατευθύνσεων. Αντιλαμβανόμαστε πως οι καταστώσεις επισφάλειας ε, συχνά οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν να λαμβάνουν. Στη Σλοβακία, παραδείγματο χάρη, έχουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο εγγυήσεων. Όπω είπε και ο συνάδελφο από το ΕΛΚ, η πρόταση αυτή είναι σωστά δομημένη, περιέχει μέτρα τα οποία θα βοηθούσαν πάρα πολύ στο να αντιμετωπίζουμε τις λεγόμενες προληπτικές αναδιαρθρώσεις και επίσης αναφέρονται και μέτρα τα οποία θα μπορούν να ε, διασώσουν θέσεις εργασίας και βεβαίως ε, καλύπτει και το ζήτημα διασυνοριακών χρεοκοπιών, ε, κάτι το οποίο εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει χρόνος και περιθώριο έλιγμων έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να βρει μία διέξοδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ε, απαιτείται άμεση δράση, κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει ε, περικοπές σε μισθούς, ε, σε μπόνους κτλ. Οπότε πολλές τροπολογίες κοιτάνε αυτό το θέμα και θεωρούμε ότι αυτές οι τροπολογίες έχουν πολύ καλές προθέσεις, αλλά θεωρούμε ότι κάποιες από αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε αντιπαραγωγικά αποτελέσματα γιατί θα καθυστερήσουν και θα σταματήσουν την διαδικασία αναδιάρθρωσης και τελικά η επιχείρηση θα κλείσει και θα χαθούν όλες οι δουλειές. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν κρίνουμε τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Σαμπών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω στη γλώσσα του Θερβάντες και, ε, και θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μαρτέν κατέχει άπτεστα αυτή τη γλώσσα, το γνωρίζω. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να σταθώ σε ζητήματα γενικού περιεχομένου. Μιλώ για την εξαιρετική εργασία της Κομισιόν και του κυρίου Μαρτέν του Ιδίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και σχετίζεται με πολλές πτυχές. Είναι ένα οριζόντιο ζήτημα. Εγώ είμαι εισηγητής της ΕΚΟΝ που ε, είναι συνυπεύθυνοι με την Γιούρη και μου είπαν ε, από την ε, πρεσβεία της Ισπανίας ότι όταν πρόκειται για μια διαδικασία συντονισμού σε εθνικό επίπεδο ασχολούνται 17 φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον για θέματα συντονισμού. Ευχαριστώ για το ότι έθεσε επιτάπητος αυτό το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή μιλάμε για τις 800.000 τους οποίους ε, προαναφέρθηκε η συνάδελφος από την Πολωνία. Μιλάμε για τις μικροεπιχειρήσεις και τις πιο ευάλωτες κατηγορίες επιχειρήσεων. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη. Οι μικροεπιχειρήσεις αργοπεθαίνουν. Γι' αυτό θα πρέπει να τους δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία να επιβιώσουν. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ή θα τις διατηρήσει. Υπάρχει το θέμα της επικουρικότητας, γιατί τα χρηματοοικονομικά συστήματα σε κάθε χώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Στο τομέα των κατασκευών στη χώρα μου υπήρχαν ορισμένες ε, στάσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια φούσκα, η οποία όταν έσπασε οδήγησε στο να ανακαλύψουμε το θνησιγενή χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτέν. Υπάρχουν και άλλες πτυχές που σχετίζονται με τα δικαιώματα των εργαζομένων. δεν δεχόμαστε να κατεβεί ο πύχης των δικαιωμάτων. Αυτό είναι απόλυτα σαφές και υπάρχει πλήρης προστασία σε νομοθετικό επίπεδο. Τώρα θα πρέπει να δράξουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή, της δεύτερης ευκαιρίας, για να βελτιώσουμε αυτά τα ε, δικαιώματα. Θα πρέπει να δούμε ε, δηλαδή τι επιπτώσεις υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Θα θέλαμε όμως να μην αργοπεθαίνουν οι επιχειρήσεις και να μην χάνονται, ε, και να μην χάνονται θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πεμπτουσία του ζητήματος. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να περιπλέκουμε άσκοπα το ε, ζήτημα. Ε, σε σχέση με τους whistleblowers, με τους ε, καταγγέλλοντες, στην ουσία ε, καταγγέλουν παράνομες δραστηριότητες. Αλλά πώς θα τους προστατεύσουμε. Και αυτό αφορά και τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να εξισορροπήσουμε την κατάσταση για την δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε επουδενή μείωση ε, ή ε, το να χαμηλώσει ο πύχης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ως προς την αρχή της επικουρικότητας, μας ενδιαφέρει η αποκέντρωση, γιατί αν πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την ουσιώδη πρωτοβουλία της δεύτερης ευκαιρίας, θα πρέπει να την εντάξουμε στο χρηματοοικονομικό πλαίσιο που τη διέπει. Δηλαδή, θα πρέπει να δεχτούμε μία οικονομική και κοινωνική συλλογιστική για να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή την ε, ευημερία των εργαζομένων εκεί όπου μπορούμε. Η Παλώμα Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτέν για την εργασία του, για την προστασία των εργαζομένων. Θα ήταν απαράδεκτο αυτή η ρύθμιση ε, να επιλύσει την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που θα απαλλαγούν από τα στοιχεία παθητικού κατά των εργαζομένων. Δεν θα δεχτούμε την κερδοσκοπία των επιχειρήσεων με βάση το μισθολογικό των εργαζομένων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν το δικαίωμα πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που όμως δεν τηρείται κατά τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το κείμενο ενισχύοντας και τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε και την έννοια των ομαδικών απολύσεων σε σχέση με την αναδιάρθρωση. Θα πρέπει να γίνουν χρηματοοικονομικές προσαρμογές για να μην παρέμβουμε με το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που έχουμε αναγνωρίσει για να μην γίνονται ε, βήματα τακτικισμού από τις επιχειρήσεις ε, όπου συγκαλύπτεται η λογιστική απάτη για να αποδυναμωθεί η θέση των εργαζομένων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εμπειρία μας ως προς τη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που είναι αφαιρέγγιες αλλά τις ανοκτούν οι εργαζόμενοι, όπως ισχύει με τους συνεταιρισμούς. Για να διατηρήσουμε την εργασία των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις όπου υπάρχει μια κατάσταση κρίσης που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει κανείς από τους πρασίνους ή από το EFTD. Ο κύριος Ντομινίκ Μαρτά, λοιπόν, έχει το λόγο για να συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να δούμε το θέμα της προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και τη διαδικασία υγιούς αναδιάρθρωσης για να αντιμετωπίσουμε την αφαιρεγγιότητα και την απαλλαγή. Το θέμα αυτό είναι πολύ σχηδές. Κατά την άποψή μας, το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Εντουάρ Μαρτά ε, περιέχει πολύ θετικές ιδέες. Είμαστε υπέρ των εναλλακτικών σχεδίων που θα προβάλλουν οι εργαζόμενοι και το δικαίωμα έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό. Θα θέλαμε ο εισηγητής να μας πει ποιες είναι οι τροπολογίες για το άρθρο 10 και ε, λυπούμεθα διότι τα μη, εξυ... μη οφειλές δεν αντιμετωπίζονται. Επίσης, οι κρατικές επιδοτήσεις δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο μίας παραγράφου μόνο στη σελίδα 13. Θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τις χρηματοοικονομικές πτυχές και την λειτουργία των hedge funds που θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υποστηρίξουμε ή όχι. Θα πρέπει να δούμε και τις κατασυρωήν πτωχεύσεις και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να πει ε, κάτι η κυρία Καρσέα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης και τους κοιόδες εισηγητές για τα σχόλια. Λίγες διευκρινήσεις να δώσω για το τι σκόπευε η Κομισιόν με αυτήν την πρόταση. Βεβαίως, σε σχέση με τους εργαζόμενους δεν θέλαμε να θίξουμε το υφιστάμενο και εκτιμένο και τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό το οποίο θέλαμε ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στις εταιρείες να αναδιοργανωθούν και να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στην διαδικασία αυτή και κοιτώντα το τι είδου εταιρείε θέλουμε να έχουμε σε αυτές τις διαδικασίες κοιτάξαμε συγκεκριμένα την τεράστια πλειοψηφία των εταιριών που είναι μικρομεσές Πάνω από το 99% των εταιριών και αυτή τη στιγμή δεν ωφελούνται από τέτοιες διαδικασίες αναδιάρθρωσης λόγω του κόστους και άλλων αντικινήτρων που ε, θεωρούν οι ιδιοκτήτες μικρών εταιριών ότι είναι δυσανάλογα. Οπότε, σε πολλά σημεία στην πρόταση προσπαθήσαμε να γίνει η διαδικασία πιο ελκυστική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό αφορά παραδείγματος χάρη προτάσεις για τη μείωση του κόστους όπως π.χ. το να μην ε, υπάρχει υποχρεωτικός ορισμός ε, μεσολαβητών ε, αφαιρεγγιότητας σε κάθε περίπτωση. Ξέρω ότι έχετε προτείνει κάποια πράγματα σχετικά. Ε, υπάρχουν πολλές τροπολογίες για την χρήση εμπειρογνωμόνων που κοστίζουν. Και για μια εταιρεία που έχει ήδη οικονομικές δυσκολίες και αντιμετωπίζει διαδικασία χρεοκοπίες θα ήταν υπερβολικό να ζητήσουμε να πληρώσει και τέτοια γνωμοδότηση ο ίδιος ο φιλέτης. Οπότε σκοπεύαμε να μειώσουμε το κόστος για τον οφηλέτη και όχι να προσθέσουμε περαιτέρω. Μετά. Αναγνωρίζουμε βεβαίως την σημασία των μέσων έγκυρης προειδοποίησης. Έχουμε το άρθρο 3, το οποίο προβλέπει κάποιες ελάχιστες αρχές όμως το εκτιμώντας 16 αναπτύσσουμε λίγο αυτό το σκεπτικό της έγκαιρης προειδοποίησης και εκεί πέρα υπάρχει ευελιξία για διάφορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη, παραδείγματο χάρη συνδικάτα ε, ή πληροφοριοδότες, όμως ε, να σκεφτήκαμε να γίνει υποχρεωτικό αυτό για όλα τα κράτη-μέλη, γνωρίζοντας ε, και τις υφιστάμενες νομικές ε, παραδόσεις. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω λοιπόν είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν κάποιες αρμοδιότητες σε εκπροσώπους εργαζομένων ή σε καταγγελούντες, αλλά δεν είναι υποχρέωση. Επίσης, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην πρότασή μας προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών. Σε κάποια κρατημέλη οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ σύντομες, τρεις-τέσσερις μήνες το πολύ, χωρίς δυνατότητα επέκταση Σε άλλα κρατημέλη είναι δυνατόν να επεκταθούν οι διαδικασίες ε, μέχρι τους 12 μήνες, 18 μήνες με συγχωρείτε, ή μέχρι και δύο χρόνια. Οπότε προσπαθήσαμε να υπάρχει βεβαιότητα για όλα τα μέρη, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να υπάρχει ένα απόλυτο όριο των 12 μηνών ως maximum, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν την ευελιξία να έχουν ακόμα πιο σύντομες διαδικασίες, όπως είπα, 3 ή 4 μήνες. Οπότε, εάν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, πολλά βήματα αυτά μπορεί να μην είναι δυνατά σύμφωνα με το εθνικό δικαίο, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση τέτοια για όλα τα κράτη-μέλη και αυτό παραδείγματο χάρη να αφορά την χρήση εμπειρογνωμόνων που συνήθως χρειάζεται χρόνο και μπορεί να είναι ασύμβατο με κάποια πιο σύντομη διαδικασία. Αυτές είναι οι γενικές μου παρατηρήσεις για την ώρα. Ευχαριστώ ε, να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε για κάτι πιο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Κύριε Μαρτάν, θέλετε να πείτε, να συμπληρώσετε κάτι. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Μόνο ορισμένα σχόλια. Δεν θα απαντήσω σε όλους. Χαίρομαι όμως διότι όλοι θέλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αποτρέψουμε τις ε, πτωχεύσεις. Φυσικά τα μέσα διαφέρουν και εγώ δεν θα ήθελα να επιβάλλω μία άποψη σε σχέση με αυτά που είπε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, θα πρέπει να βασιστούμε στα ε, ήθη και έθιμα της εθνικής νομοθεσίας, αλλά νομίζω ότι υπάρχει το δικαίωμα της πραγματογνωμοσύνης και το δικαίωμα πραγματογνωμοσύνης στη Γαλλία αφορά επιχειρήσεις ενός μεγέθους και άνω, δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 50 εργαζόμενους δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, τουλάχιστον στο δικό μας εθνικό δίκαιο. Εάν δούμε τώρα ποιες είναι οι χώρες που βρίσκονται σε καλύτερη θέση, στρέφουμε τα βλέμματά μας προς τη Γερμανία, γιατί υπάρχει ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος εκεί και οι διαπραγματεύσεις ε, είναι ένα δικαίωμα το οποίο θα μπορούσα να πω ότι είναι τόσο θεσμοθετημένο που είναι σαν να έχει ένα γενετικό κώδικα. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να λάβουμε υπόψη ότι και τα συνδικάτα δέχτηκαν να κάνουν υποχωρήσεις αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι και η νομοθεσία προσαρμόστηκε ε, σε αυτές τις προσπάθειες που έκαναν οι εργαζόμενοι. Στη Γερμανία δηλαδή υπάρχει δικαίωμα μερικής ανεργίας που επεκτάθηκε στους 24 μήνες έτσι ώστε να αποφύγουμε πτωχεύσεις Πιστεύουμε λοιπόν ότι για να αποφύγουμε ακραίες καταστάσεις θα πρέπει να γίνονται διαπραγματεύσεις. Δηλαδή οι μισθωτοί καταβάλουν συνήθως ε, προσπάθειες για να περισωθούν τα πράγματα και για να αποσοβηθεί μία μεγάλη κρίση και οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση επιχείρησης και θα ειδοποιήσουν ε, όταν ε, η κατάσταση δεν πάει καλά. Παρακολουθώ δεκάδες επιχειρήσεις και όχι μόνο στη Γαλλία όπου οι εργαζόμενοι ειδοποιούν για την κατάσταση αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ολοένα και χαμηλότερη δυνατότητα πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης. Δηλαδή, ε, δυστυχώς όταν συνταξιοδοτείται κάποιος, προσλαμβάνεται κάποιος άλλος, αλλά έχει ένα καθεστώς ε, ορισμένου χρόνου αποκλειστικά. Άρα θα πρέπει να προωθήσουμε τις συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο. Δημιουργούν πλούτο. Δεν λέμε ότι τα συνδικάτα θα, θα πάρουν την εξουσία στις επιχειρήσεις. Απλώς λέμε πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να βοηθήσουν έτσι ώστε να ορθοποδήσει μια επιχείρηση γιατί σίγουρα και οι εργαζόμενοι είναι μία σοβαρή πηγή πληροφορίας και μπορούν να προβούν σε μία σωστή διαπραγμάτευση, δηλαδή κατέχοντας τα στοιχεία που πρέπει για να αποσοβήσουμε κινδύνους και ιδιαίτερα την πτώχευση. Έτσι δίνουμε μία δεύτερη ευκαιρία. Ξέρουμε και έχουμε πολλαπλά παραδείγματα όπου είχαμε οργανωμένες πτωχεύσεις από την μητρική. Δείτε τι έγινε στο Βέλγιο με την κατερπίλαρ. Οι εμπειρογνώμονες έδειξαν ότι η πτώχευση ήταν προοργανωμένη από την μητρική εταιρεία. Μιλώ για την πτώχευση της Caterpillar στο Σαρλερουά. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει σωστή πραγματογνωμοσύνη. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει μία θεμητή διαπραγμάτευση και δεν θα υπάρχει το ίδιο επίπεδο γνώσης του αντικειμένου. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, προειδοποίηση που μπορούν να προβάλλουν μόνο οι εργαζόμενοι. Άρα χρειάζεται να προστρέξουμε στην ε, πηγή της ε, πληροφορίας και γι' αυτό υπάρχει και το δικαίωμα πραγματογνωμοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ και κατέγραψα όλα σας τα σχόλια, τα οποία θα λάβω σοβαρά υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία η 10η Μαΐου στις 12, προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Α, με συγχωρείτε, 17 Μαΐου. Είπατε να παρατείνουμε 17 Μαΐου. Ήταν η 10η Μαΐου, αλλά επειδή η Γιούρη χρειάζεται χρόνο, Έχουμε περιθώρια και θα ε, σας έλεγα να παρατείνουμε μέχρι τις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, αν συμφωνείτε όλοι. Καμία αντίρρηση. 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι και θα εγκρίνουμε στις 12 Ιουλίου στην Επιτροπή Απασχόλησης και η Γιούρη θα ψηφίσει το Νοέμβριο, 20-21 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Ε, αν δεν έχετε κάτι να θίξετε, κάτι το διαφορετικό, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 29 και 30 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ. Γεια σας.